Νοεμβρίου 2014 ε, εξετάστηκε ε, το αίτημα των αρχών της Ρουμανίας για τον κύριο Νίκα για την άρση ασυλία του. Σύμφωνα με τον κανονισμό διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων η οποία και